So, Κυρίες και κύριοι, ας συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. Θα περάσουμε τώρα στο σημείο 13. Τελευταίο σημείο, παρουσίαση μελέτης σχετικά με τις επιπτώσεις προστατευτισμού στη διεθνή διπλωματία. Πρόκειται για μια κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου. Θα ήθελα να καλωσορίσω τα μέλη της ΣΥΝΤΑ και ιδίω τον Προεδρό μας, τον κύριο Λάγκε. Τώρα, η μελέτη ζητήθηκε από τις Επιτροπές ΑΦΕΤ και ΙΝΤΑ πέρσι τον Ιούνιο και δεν χρειάζεται να τονίσω τις ε, τάχεις εξελίξεις στον τομέα του τελευταίους μήνες. Επίσης ενημερώθηκα ότι ο εμπειρογνώμονας μας έπρεπε να επικαιροποιήσει το κείμενο πολλές φορές προκειμένου να συμπεριλάβει νέα γεγονότα. Θα ήθελα να καλωσορίσω την εμπειρογνώμονά μας, την κυρία Καμαλατεουάρ, η οποία είναι ειδικό ε, σε διεθνέ και ευρωπαϊκό εμπορικό δίκαιο, στι δημόσιε συμβάσει, στον ανταγωνισμό και στην ε, πολιτική καταναλωτών. Έχει διδακτορικό στο Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο της Γενέβης, ε, έχει μεταπτυχιακό στο Διεθνό και Ευρωπαϊκό Εμπορικό Δίκαιο από το Πανεπιστήμιο του Άμστερνταμ. Ε, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην εμπειρογνώμονά μας, αν μπορείτε να μας μιλήσετε για 15 λεπτά περίπου και μετά θα έχουμε χρόνο για τη συζήτηση. σας ευχαριστούμε που ήρθατε από το Άμστερνταμ στις Βρυξέλλες. Σας ευχαριστώ που με καλέσατε είναι πραγματικά μου να βρίσκουμε εδώ και να υλοποιήσω την έκθεση. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη ένταση και αστάθεια στις διεθνείς υποθέσεις ε, και με βοήθησε όλα αυτά να τα δω με ένα συστηματικό τρόπο. Το βασικό μήνυμα από όλη την έκθεση είναι ότι υπάρχουν πολλές προκλήσεις ε, ε, στην συνένεση που οικοδομήθηκε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο Πολύ μεγαλώσαμε και πιστεύουμε ότι αποτελούσε την ασφαλεία μας, αλλά επίσης υπάρχει και λύθη. Ξεχνάμε γιατί ε, οικοδομήθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε ειρήνη μέσω του εμπορίου. Αυτά τα θέματα προέκυψαν ε, στα διάφορα κεφάλαια και άλλο ένα θέμα που ανέκυψε ήταν ε, ότι στην εξωτερική πολιτική εισέρχεται πλέον και το διεθνές εμπόριο. Θα σα ε, παρουσιάσω μια επισκόπηση τη εκθεση. Είχαμε ένα κεφάλαιο για το γύρο τη Τόχα και τον ΠΟΕ και περάσαμε στη στάση των ε, Ηνωμένων Πολιτειών και την ε, παραδοσιακή στάση τους καθόπιν για τον Brexit. Επίσης, πώς θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να θασέψει την παγκοσμιοποίηση και το τελευταίο κεφάλαιο αφορούσε την Κίνα και τις απειλές της Κίνας πριν τα γεωπολιτικά συμπεράσματα. Θα σας παρουσιάσω το κεφάλαιο εν συντομία και ελπίζω ότι μπορούμε να έχουμε μια συζήτηση ενδιαφέρουσα στη συνέχεια. Πολυμερισμός στο εμπορίο ΠΟΕ είναι ο πιο ισχυρό ε, διεθνής οργανισμός ε, με έναν ε, μηχανισμό δεσμευτικό για την διευθέτηση, για την επιλύση των διαφορών. Δυστυχώς αυτό που έγινε υπό το γύρο της Δόχα είναι ότι υπήρξε ε, μια ε, διαφωνία μεταξύ των αναπτυσσόμενων και των αναπτυγμένων χωρών, γιατί από ό,τι φαίνεται οι αναπτυσσόμενε χώρε φαίνεται να ζητούν περισσότερε παραχωρήσει από τι αναπτυγμένε χώρε, κυρίω στο θέμα τη γεωργία. Και αυτό οδήγησε σε αδιέξοδο. Ξεκίνησε το 2001 ο γύρο τη Ντόχα και όταν ξεκίνησε ήμασταν ε, ουσιαστικά υπό την απειλή τη τρομοκρατία και υπήρχε μεγάλη βούληση στην Ντόχα που δεν συνεχίστηκε από τότε. Αυτό που ακούσαμε είναι ότι υπήρχε ένα ε, πρόβλημα με την εννέα επιχείρηση, είναι ότι ε, προχωράμε ε, σε όλα τα θέματα και όχι σε υποτομιακή βάση. Και μπορείτε να φανταστείτε ότι υπήρξε ένας μηχανισμός συνένεσης και έπρεπε να συμφωνήσουν σε όλα. Επομένως δεν συνέβησαν πολλά από το 2001 και φτάσαμε στο σημείο να ρωτιούνται διάφορα τι ακριβώς κάνει ο ΠΟΕ επειδή το νομοθετικό σκέλος ε, του ΠΟΕ ε, έχει τελματώσει, έχει ουσιαστικά επιβαρυνθεί το δικαστικό σκέλος του ΠΟΕ και τώρα τους ε, κατηγορούν για δικαστικό ακτιβισμό και αυτό προκαλεί σύγχυση σε μέρη όπως οι Ηνωμένε Πολιτείε. Έτσι λοιπόν, όταν πρόκειται για διορισμό ανθρώπων ε, για το ανώτατο ε, σώμα, ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν θέσει βέτο στους διορισμούς. Έχουμε λοιπόν τρία μέλη που έχουν κατέβει, που έχουν αποχωρήσει και είναι μεγαλύτερο το άχθος. Και το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει φορέας εφέσεων, τότε ε, δεν μπορούν ε, να εκδικαστούν γρήγορα οι εφέσει και τα μέλη ή μπορεί να χρησιμοποιήσουν μηχανισμού εμπορικής άμυνας ή μπορεί να έχουν άλλους εμπορικούς πολέμους εκτός ε, του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα καθώ οι Ηνωμένε Πολιτείε υποσκάπτουν τον οργανισμό έχει υποσύρει οι ΗΠΑ την υποστήριξή τους από τον ΠΟΕ de facto και αυτό οδηγεί άλλα μέλη να αναζητούν άλλα φόρα. Ε, Παραδείγματο χάρη προσπαθούν ε, να αναζητήσουν άλλα φόρα όπως η G20 και η G7 και αυτό υποσκάπτει τον ΠΟΕ. Έτσι λοιπόν... Ε, αυτό που ήταν ένας ισχυρός διεθνής οργανισμός υποσκάπτεται. Και φυσικά οι αναπτυσσόμενες χώρες έχουν μεγάλο πρόβλημα με την εντολή του ΠΟΕ, αλλά φυσικά αυτό δεν είναι τόσο επικίνδυνο όσο η απόσυρση της υποστήριξης των ΗΠΑ, σε ό,τι αφορά το ρόλο των ΗΠΑ. Ε, οι Ηνωμένε Πολιτείε τα τελευταία 50 χρόνια ήταν ηγέτης σε ηγετική θέση στο διεθνές ε, σύστημα μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο είχαμε τον ψυχρό πόλεμο. Οι Ηνωμένε Πολιτείε χρειάζονταν την διεθνή κοινωνία και χρειάζονταν συμμάχου ε, για να αντιταχθούν ε, στην ε, Ρωσία. Όμω μετά το 1995 δεν χρειάζονταν πλέον αυτού του συμμάχους γιατί κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση και τώρα οι Ηνωμένε Πολιτείε είναι ο αντιαφισβήτητος ηγέτης σε οικονομικό και στρατιωτικό επίπεδο και από τον Τόναλτ Τραμπ βλέπουμε ότι μπορούν να αγνοούν τη διεθνή κοινότητα και να υποστηρίζουν να αποσύρουν συγγνώμη, την υποστήριξη για τη διεθνή αρχιτεκτονική χωρίς ιδιαίτερε δυσκολίε. Έχουν αποσύρει λοιπόν την υποστήριξή τους. Και τώρα μπορούμε να μιλήσουμε για ε, ε, ουσιαστικά μία ε, διαδικασία διάλυσης, προληπτικής διάλυσης δημιουργίας άλλων σχηματισμών και μπορούμε να το δούμε αυτό στο γεγονός ότι πολλές χώρες δεν ξέρουν ποιε είναι οι φιλοδοξίε των ΗΠΑ, πέρα από το America First, η Αμερική πρώτα, και δεν ξέρουν τι συμβαίνει στη διεθνή κοινωνία, απλώ ξέρουν ότι δέχονται απειλέ. Και επειδή οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, αποσύρονται από πολλές πολυμερείς και διμερείς διαπραγματεύσεις, έχουμε τώρα μία ε, περίεργη διμερή συζήτηση με το Μεξικό που αποκλείει την Κίνα, έχει αποσυρθεί από την TTIP, οι Πολιτείε και από την TTP και αυτό δημιουργεί ένα κενό εξουσία, το οποίο είναι πιο εμφανέ στην περιοχή Ασία Ειρηνικού. Αυτό επέτρεψε στην Ασία να εισέλθει ε, στο προσκήνιο. Αυτό προκαλεί αποσταθεροποίηση γιατί η Κίνα είναι νέο παίκτη σε διεθνέ επίπεδο. Και φυσικά προκαλεί ανησυχίε ε, σε άλλου όπω η Ιαπωνία. Έτσι λοιπόν αποσύρεται από το τον ε, και έτσι συνεισφέρει στην αποσταθεροποίηση. Όμως ε, μπορεί ακριβώς, ε, αυτή μπορεί να είναι η πολιτική των είπα αυτή τη στιγμή, η αποσταθεροποίηση. Το όραμα του Ηνωμένου Βασιλείου, άλλη επιλή οικονομικού εθνικισμού. Μπορείτε να δείτε ότι πρόκειται για μια επίθεση κατά της παγκοσμιοποίησης. Πολλοί άνθρωποι ένιωθαν ότι είναι στο περιθώριο όμως ε, ο λαϊκισμός ε, καλλιεργείται μέσω του Brexit επιτυχώς στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι πολιτικοί μπόρεσαν να κατηγορήσουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και την παγκοσμιοποίηση για ορισμένους τομείς που στο Ηνωμένο Βασίλειο, ε, όπου στο Ηνωμένο Βασίλειο είχε σημειωθεί αποτυχία των δημοσίων πολιτικών. Είχαμε πολλά προβλήματα που δεν είχαν να κάνουν την Ευρωπαϊκή αλλά πρόκειται για ε, χώριες πολιτικές έτσι λοιπόν η ψήφος για τον Brexit αποτέλεσε σοκ για όλους, ακόμη και για όσους ε, ψήφισαν υπέρ του Brexit. Τώρα υπάρχουν κάποιες κόκκινες γραμμές που θα καθορίσουν το ρόλο της Βρετανίας εκτός της Ένωσης. Έτσι λοιπόν η μετανάστευση και η κυριαρχία είναι μεγάλες κόκκινες γραμμές. Αυτό δημιουργεί επιλογές και μη επιλογές, μια μη επιλογή. Αν ε, ε, διατηρήσουμε ε, το εργατικό θέμα εκτός ε, των σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Παίρνουμε το χάρη δεν είναι ανοιχτό το μοντέλο του ΕΟΧ, το μοντέλο της ΕΣΕΣ με τη ΣΕΝΚΕΝ δεν είναι ανοιχτό. Έτσι λοιπόν τι θέλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Μπορεί να έχει μια καλλιτελωνιακή ένωση με το Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά είδαμε ότι η τελωνική ένωση με την Τουρκία δεν ήταν πολύ επιτυχής. Έχουμε τώρα ηλεκτρονικό εμπόριο. Έτσι λοιπόν ε, δεν ξέρω αν θα ήταν, μια πολύ, ενδια... θα πολύ ενδιαφέρουσα μια τέτοια τελωνιακή ε, ζώνη και ζώνη αγαθών. Ε, για το Ενωμένο Βασίλειο λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να επαναφεύρει τον τροχό. Πολύ πολιτική είναι κατά της ιδέας αυτής ότι ε, θα υπάρχει ε, σημαντική επίπτωση στο εμπόριο από την πρώτη μέρα. Αλλά αυτή είναι μία από τις λίγες εναλλακτικές που έχουμε αν, διατηρήσουμε τις κόκκινες γραμμές στη μετανάστευση. Έχουμε λοιπόν πρόβλημα στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπάρχει έλλειψη οράματος για το μέλλον και έλλειψη τρόπων να φτάσουμε σε αυτό το όραμα, οδών να φτάσουμε σε αυτό το όραμα και είναι κάτι λυπηρό αυτή τη στιγμή στο Ηνωμένο Τώρα, το όραμα τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει πρόβλημα η Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί εξωτερικά χρειάζεται τις περιφερειακές Εμπορικέ Συμφωνίε και την παγκοσμιοποίηση. περισσότερη ανάπτυξη είναι εκτό τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει διεθνεί γέφυρε όμω εσωτερικά η ίδια απογοήτευση που υπάρχει στο Ηνωμένο Βασίλειο και στη ΣΥΠΑ και πολλέ ε, χώρε. Ε, κυριαρχεί και αποτελεί παναχώρηση. Έτσι λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να χαλιναγωγήσει αυτές τις δύο διαφορετικές δυναμικές ε, και φυσικά το Brexit αποτελεί οικονομική απώλεια, αλλά αλλάζει και την ισορροπία της ε, εξουσίας. Εσωτερικά η Ευρωπαϊκή Ένωση αντιμετωπίζει νέους ε, ανασχηματισμούς, μπορεί η αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου να επιτρέψει πιο συγκεντρωτικές πολιτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς ε, τον μπλοκ ε, των Βρετανών που χαράσουν πολιτικές, ε, όμως και πάλι χάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε συνεισφορά και αναφερόμαστε στην έκθεση στο τι συμβαίνει στην δυναμική ε, τη ψηφοφορία τη Ευρωπαϊκή Ένωση, τη ψήφου τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθεί λοιπόν να αντιθασέψει η Ευρωπαϊκή Ένωση την παγκοσμιοποίηση και να παρουσιάσει ένα όραμα για το πώ μπορεί η παγκοσμιοποίηση να βοηθήσει του ανθρώπου, ε, προκειμένου να μπορούν να υποστηρίζουν οι άνθρωποι τι ε, εμπορικέ συμφωνίε. Είναι όμω δύσκολο γιατί πολλοί άνθρωποι θεωρούν ότι η παγκοσμιοποίηση δεν του έχει βοηθήσει. Τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει το ταμείο της επεξημοποίησης, ε, όπως και άλλα μέσα, μέσω των οποίων αποζημιώνει ε, αυτούς που χάνουν. Όμως, ε, ίσως να μην έχουν χρησιμοποιηθεί πλήρως αυτά τα εργαλεία. Το Ηνωμένο Βασίλειο Χάρη δεν έχει χρησιμοποιήσει αυτό το ταμείο. Υπάρχει έλλειψη λοιπόν επικοινωνίας σε σχέση με τους μηχανισμούς που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους απλούς πολίτες. Και φυσικά αυτό υποσκάπτει την ικανότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, να βγει και να διαπραγματευτεί από μια ισχυρή θέση τις εμπορικές συμφωνίες. Ε, είδαμε και τα κινήματα, σταματήστε την TTIP κτλ. Στο επόμενο κεφάλαιο ήταν η Κίνα. Η Κίνα είναι ενδιαφέρουσα γιατί έχει ε, μεταμορφωθεί τις δύο τελευταίες δεκαετίες και φαίνεται να είναι υπέρ της παγκοσμιοποίησης. Η ηγεσία υποστηρίζει τον ΠΟΕ και ε, καταδικάζει τις ε, παραβιάσεις του πολυμερούς εμπορικού συστήματος. Ταυτόχρονα όμως ξέρουμε ότι η Κίνα εξακολουθεί να επιδιώκει τον σοσιαλισμό με κινέζικη, ε, στην κινέζικη του εκδοχή. Και ενώ πιστεύουμε ότι η Κίνα απειλή τη Η Κίνα έχει πολλά εσωτερικά προβλήματα εσωτερικά με ανισότητα, φτώχεια, εθνίκε συγκρούσει. Τι προσπαθεί να κάνει η Κίνα. Έχει αυτή την πολιτική, μια ζώνη, μια οδό. θέλει να επενδύσει στου γειτονέ τη και να οικοδομήσει τις, εθν... τις ε, διεθνείς της σχέσεις. Όμως ε, ξέρουμε από δηλώσεις από χώρες όπως η Μαλαισία υπάρχουν ε, προβλήματα με τις επενδύσεις της Κίνας υπό τον πρωτηλή αυτή. όλα αυτά τα θέματα τα οποία αφορούν την ανησυχία Ευρωπαϊκή Ένωση ε, παραδείγματος χάρη τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα περιβαλλοντικά ζητήματα, ε, αμφισβητούνται υπό την πολιτική μία ζώνη, μία οδός. Και αν οι Κινέζοι θεωρήσουν ότι δεν επωφελούνται από, παρά τις θυσίες, ε, τότε θα υπάρχει οπισθοδρόμηση και εντό της Κίνας και θα πρέπει να το επιλύσουν αυτό οι ηγέτες αν θέλουν να διατηρήσουν τη σταθερότητα εντό της Κίνας. Έτσι λοιπόν οι δράσεις της Κίνα απειλούν ε, τη γεωπολιτική σταθερότητα της περιοχής αλλά και παγκοσμίω, γιατί μετακινούν το κενό που έχουν αφήσει πίσω οι ΗΠΑ. και επίση η Κίνα συμμετέχει στην πολιτική 16 συνένωση στην Ευρώπη. Ε, δηλαδή ε, μπαίνει σε ευρωπαϊκές χώρες και τους προσφέρει διάφορα είδη επενδύσεων αλλά αμφισβητείται αν υπάρχει ε, ουσιαστικά επιδότηση από την κινέζικη κυβέρνηση και υπάρχει και αμφιβολία για το αν γίνονται σεβαστές οι απαιτήσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι λοιπόν, αν ε, κάποιες από τις ανατολικές ε, χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, δουν ότι έχουν καλύτερη συνεργασία με την Κίνα παρά την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Έχουμε λοιπόν αυτές τις εντάσεις σε διάφορα μέρη του κόσμου και φαίνεται σαν κάποια χρόνια μετά από την εφορία του τέλους του ψυχρού πολέμου που όλοι μιλούσαν για τη φιλελεύθερη δημοκρατία φαίνεται σαν να μην ισχύουν όλα αυτά, σαν να μην αληθεύουν. Οι κυβερνήσεις δεν ξέρουν πώς ακριβώς να αντιμετωπίσουν τις εξωτερικές και εσωτερικές πιέσεις. Θα κλείσω λοιπόν την παρουσίασή μου γιατί μπορούμε να τα συζητήσουμε τα υπόλοιπα στις ερώτα απαντήσεις. Ξεχνάμε την ιστορία, είναι σαφές, ξεχνάμε γιατί εμπορευόμαστε και τι συμβαίνει όταν έχουμε προστατευτισμό και έχουμε εμπορικούς κανόνες και φυσικά εν μέρη αυτό είναι γενολογικό αλλά αποτελεί εν μέρη και απουσία, ε, μάλλον αποτυχία των κυβερνήσεων να διαβιβάσουν το μήνυμα. Ε, δεν έχουν διαβάσει το μήνυμα πόσο έχει μειωθεί η ανέχεια ε, μέσω του εμπορίου. Όλα αυτά τα διδάγματα φαίνεται να έχουν χαθεί λόγω του ότι ο οικονομικός ε, νασιοναλισμός ισχυρή φωνή σήμερα. Έτσι λοιπόν, ε, θα ήθελα να σας πω ότι χάρηκα πολύ που συνέταξε την εκθεσία αυτή και αναμένω τις ερωτήσεις σας. Thanks a lot. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ χρήσιμη περιγραφή της κατάστασης, αλλά τώρα είναι σειρά μας να αντλήσουμε τα συμπεράσματα. Ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Ο λόγος στον κύριο Παντσέρη. Ευχαριστώ. Έχω δύο ερωτήσεις. Σε σχέση με την παρουσίασή σας. Η πρώτη ερώτηση είναι εξή. Θέλω να ρωτήσω αν εμείς, σύμφωνα με τα όσα μας είπατε. Βλέπουμε την απέτηση να καλυφθεί ένα κενό. Μα ακούτε? Όχι. Okay. Εσεί Εσείς είπατε ουσιαστικά ότι η Κίνα κάλυψε ένα κενό που άφησαν οι Ηνωμένε Πολιτείε στην παγκόσμια αγορά. Αυτό φαίνεται να αποτελεί μία πρόσκληση στην Ευρώπη να ξαναλάβει μία πρωταγωνιστική θέση στην εμπορική πολιτική. Αναρωτιέμαι αν βιώνουμε απλώς ε, μια, ένα αίτημα τεχνικού χαρακτήρα ή αν αντίθετα είμαστε σε μια στιγμή όπου χρειάζεται να προσφέρουμε και μια ποιότητα στη διαδικασία της διεθνούς εμπορικής πολιτικής. Γιατί οι ανησυχίες που μας παρουσιάσατε ε, συνέπειες που παρουσιάστηκαν από το εμπόριο και ήταν δύσκολο να τις διαχειριστούμε, θα έχουμε επανάληψη αυτής της διαδικασίας αν δεν εισαγάγουμε και την ποιοτική διάσταση. Πριν λίγο κάναμε μια συζήτηση στην επιτροπή αυτή με τον ε, νεοδιοριστέντα πρέσβη στην Κίνα. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, γιατί δεν μιλάμε μόνο για την ε, εμπορική πολιτική, αλλά και ε, υπάρχει και το πρόβλημα της ε, πολιτικής επενδύσεων που ακολουθεί η Κίνα στην Αφρική. Και εδώ μιλάμε ουσιαστικά για εφαρμογή των γεών. Γιατί δημιουργούν μεταναστευτικά προβλήματα. Πώς μπορούμε εμείς λοιπόν να ρυθμίσουμε αυτή τη σύραξη ή να μπορέσουμε να συγκλίνουμε με την Κίνα για να μπορέσουμε να διαχειριστούμε καλύτερα τα προβλήματα που έχει η Ευρώπη. Uh, δύο λεπτά, δύο λεπτά χρόνος ομιλίας. Ο κύριος Ρούμπικ είναι επόμενος. Ευχαριστώ. Πολύ ενδιαφέροντα αυτά που μας παρουσιάσετε για εμάς ως κοινοβούλιο. Ε, μας ενδιαφέρει πώς βλέπετε το ρόλο της κοινοβουλευτικής συνδόδου η οποία ιδρύθηκε το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο μαζί με τον Οργανισμό Διεθνών Κοινοβουλίων έγινε μια σύνοδος στο Buenos Aires όπου συνήλθαν 300-400 βουλευτές. Είναι μια εξέλιξη αυτή, μπορεί η, η δημοκρατική πολιτική να βοηθήσει. Και το άλλο το ερώτημα είναι πώς πιστεύετε ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να υποστηρίξει καλύτερα και οικονομικά τι θα γίνει με τις εργασίες στην Ευρώπη αν συνεχιστεί αυτή η προτεξιονιστική στάση. Είναι κάτι που δεν το θέλουμε. Χέλμουτ ε, Σόλτ. Ευχαριστώ. Θέλω και εγώ να ευχαριστήσω για την μελέτη. Ένα ερώτημα. Στην εισηγήτρια. κάνουμε λόγο για τις οικονομικές στρατηγικές μέσω των πολιτικών παραγόντων και πώς θα βρούμε μια διέξοδο ε, σε αυτή την αλληλεξάρτηση που υπάρχει. Η ερώτηση είναι ο προδοξιονισμός που προωθεί ο Τραμπ είναι μήπως μία άλλη μορφή προσπάθειας επιβολής ισχύω. για να μπορέσει να θέσει νέους όρους θα μπορούσαμε να τα μελετήσουμε ανατμήματα ή αναχώρα και να δούμε τι μπορεί να κάνει η διπλωματία. Μια λογική οικονομική διπλωματία να θεματοποιήσει τις διαφορές ώστε να υπάρξει μια επικοδομητική συνέχεια και να λάβει τα μέτρα, τα κατάλληλα, στα αρμόδιες δομές και να βρει λύσεις. Ευχαριστώ, Ανελίτς. Ευχαριστώ για τη μελέτη και την προσέγγιση αυτή που μας παρουσιάσατε. Είχαμε τον πρέσβη προηγουμένως και συζητήσαμε ε, για το 6 συν 1. Θα ήθελα να σας ρωτήσω για την 16 ε, 1, συγγνώμη, κυβερνοασφάλεια. Τι ισχύει για τις αφρικανικές χώρες αλλά και για την Ευρώπη όσον αφορά την εσωτερική ασφάλεια. Βλέπουμε την κυβερνοασφάλεια στη Γερμανία η φαρπαγή δεδομένων από την Κίνα είναι πολύ μεγάλη. Και παράλληλα έχω ακόμα μια ερώτηση για το εμπόριο και την Κίνα. Στην ηλιακή βιομηχανία και ενώσιμες πηγές, υπήρχε μια συνεργασία μεταξύ Ανατολικής Γερμανία και Κίνας. Είναι ένας ε, τομέας στον οποίο υπάρχει ε, δυνατότητα εμπορίου. Το θέμα είναι οι βιώσιμοι στόχοι και πώς μπορούμε να συνεργαστούμε. Είμαστε ανεξάρτητες προς την βιώσιμη ενέργεια σε σχέση με την Κίνα που άσχει όλο και περισσότερη περιοχή στον τομέα της ολικής ενέργειας επίσης. Τι θα συμβεί την Αφρική, πώς μπορούμε να το προωθήσουμε αυτό περαιτέρω. Uh, thank you very um, Ευχαριστώ. Υπάρχουν πολλά πράγματα που δεν καλύψατε, δεν αναφέρατε. Την Ευρωπαϊκή, τον Ευρωπαϊκό Προστατευτισμό στον ε, γεωργικό τομέα και στο πλαίσιο του κύκλου της Δόχα. Το ρόλο του δολαρίου με το οποίο ελέγχει το Διεθνές Τραπεζικό Σύστημα είπατε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε ε, ψήφισαν ενάντια στο TTIP. Ίσως δεν το έκανα, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο ψήφισε ενάντια στο TTIP. Αναφέρατε χαμηλή ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υψηλή φόρη, χαμηλή ανάπτυξη και ιδιαίτερα στη Γερμανία. Δεν τα αναφέρατε αυτά. Δεν αναφέρατε το εμπορικό πλεόνασμα της Γερμανίας. Στην Κίνα έχει πλεόνασμα σε αγαθά 375 δισεκατομμυρίων με τη ΣΥΠΑ και κάτι αντίστοιχο με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν το αναφέρεται. Είναι βιώσιμο ή δεν είναι βιώσιμο. Είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Και επίση θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και το θέμα τη κλοπή πνευματικών δικαιωμάτων που γίνεται από την Κίνα όσον αφορά το Brexit. Αναφέρεται και είναι ενδιαφέρον ότι υπάρχει ίση μετανάστευση στην Ιταλία όπως και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτή είναι μία εργασία ε, που θα την έκανε ένας ε, προπτυχιακός φοιτητής. Δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε για μια τέτοια μελέτη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για μια ακόμη φορά Διαφωνώ με τον προλαλή. Μένα μου άρεσε η έκθεση αυτή. Νομίζω ότι παρουσιάζει μια καθολική πτυχή όλων των θεμελιώδων φαινομένων που πλήττουν ε, τη νέα παγκοσμία οικονομική τάξη. Φυσικά δεν μπορούμε να εμβαθύνουμε σε κάθε πτυχή. Όμως εγώ πιστεύω ότι είναι καλή η έκθεση. Θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο. Αυτό που δεν μας είπατε είναι Ποια κατά την άποψή σας θεωρείτε ότι θα έπρεπε να είναι η βέλτιστη στρατηγική που θα έπρεπε να ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσει να έχει πραγματική ηγετική θέση στο να ξαναθέσει τις βάσεις της νέας παγκοσμίας τάξης ή να συνεχίσει με μια νέα παγκοσμία τάξη βάσει Έτσι λοιπόν, ποια θα ήταν η βέλτιστη στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεύτερον. Εσείς από τη μελέτη συμπεραίνετε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική αν εγκαταλείψουν οι τον ΠΟΕ. Δύο ερωτήσεις. Πιστεύετε ότι αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να διαβαστεί στι ΗΠΑ που θεωρούν ότι όλοι εξαρτώνται από το αν υπάρχουν ή όχι. Έτσι λοιπόν συνεχίζει να δρά μέσα σε αυτή την αλαζονία. Δεν θα ήταν καλύτερο να θέσουμε ότι πράγματι υπάρχουν εναλλακτικέ και ότι μπορούμε να εργαστούμε ε, στο να βρούμε εναλλακτικέ ε, σε διεθνέ επίπεδο. Φυσικά ε, είναι μια χώρα κλειδί πολιτείες, αλλά εγώ νομίζω ότι ένα από τα προβλήματα της ε, κυβέρνησης Τραμπ είναι η προσωπικότητα του Τραμπ. Και τέλος, πώς πλήττει την Ένωση και τη συνεργασία στην Ευρωπαϊκή Ένωση το σχέδιο 16 1 με την Κίνα. Μήπως ε, ουσιαστικά πρόκειται για ένα μηχανισμό που διαρρεί την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριος, κύριος Θα ήθελα να συμφωνήσω με τον γειτονά μου δίπλα. Είπα αυτό που θέλω να πω. Είναι σαν μια κατηγορία στον υπόλοιπο κόσμο που δεν θέλει να έχει εμπορικές αλληλίες με την Ευρώπη, με τους δικούς της όρους. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας οργανισμός ο οποίος ε, καθορίζει τι θα κάνει στην επικράτειά της με τους δικούς της όρους και είναι δύσκολο να βρούμε καθαρή ε, συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ζητάει, απαιτεί από τους εταίρους να προσαρμοστούν στο δικό της τρόπο σκέψης ε, με παράλογους κανόνες να δώσει προνόμια σε άτομα, σε ομάδες όπως είναι οι γυναίκες, σε ομοφυλόφιλοι κτλ. Θέματα που θα πρέπει να έχουν θέση σε εμπορικά ζητήματα. Παράλογη στάση από την Επιτροπή που κάνουν λόγο για ελεύθερο εμπόριο, αλλά το οποίο το υποβάλλουν στις ιδεολογίες ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θεωρώ λοιπόν ότι ένα βασικό παράδειγμα αυτής της άρρωστης πολιτικής είναι η γεωργία, όπου έχουμε όρους ε, τύπου Σοβιετικής Ένωσης, όπου οι χώρες δεν μπορούν να ε, έχουν εμπορικές συναλλαγές με κανέναν άλλον πέρα από εμάς και χρειάζονται εκατοντάδες εκατομμυρίων ευρώ βοήθεια στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Κάποιοι επιστήμονες ανέφεραν ότι η Κίνα έχει ιδεολογικά στοιχεία στρατηγική τους. Ο κύριος Σούστα στη συνέχεια. Ευχαριστώ. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα. Όταν θέλουμε να σχεδιάσουμε την πολιτική όσον αφορά την ε, μελέτη. Δεν την ε, διάβασα καλά. Αλλά το ερώτημα πρώτα ε, ή όχι, το θεωρώ ελλειπές. Υπάρχουν ε, αντιφάσεις. Ο τρόπος περιγραφτεί της είπα. Φυσικά πάνω στην κοινωνία των ΗΠΑ βασίστηκε ε, το εμπόριο και αυτό σημαίνει ότι ε, κρατάει αυτό το προνόμιο το κρατάει αυτό το προνόμιο οι ΙΠΑ και θέλουν να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία πίεση που μπορούν να έχουν. Αυτό δεν μπορούμε να το πούμε για την Κίνα. Τελευταία, το Κομμουνιστικό Κόμμα στη συνέλευση ε, δήλωσαν ότι θέλουν να είναι οι πιο ισχυροί οικονομικά μέσα στα επόμενα χρόνια και για να το πετύχουν αυτό θα χρησιμοποιήσουν στοιχεία εξαναγκασμού Αν συμβεί αυτό, θα έχουμε μια μεγάλη μακροχρόνια κρίση που θα φέρει πολλά προβλήματα. Αυτό που γίνεται από την πλευρά μας είναι να κλείσουμε τη μία εμπορική συμφωνία μετά την άλλη. Ε, έχουμε αυτή την απόγνωση και αυτό δεν βοηθάει. Δεν θα πρέπει να κινούμαστε επίσης στη σκιά τον ΗΠΑ. Κάτι που το κάναμε πολύ στα χρόνια που ακολούθησαν τον ε, Δεύτερο Παγκόσμιο, Παγκόσμιο Πόλεμο. Ευχαριστώ πολύ από την πλευρά μου. Να αναφερθώ στις τελευταίες εξελίξεις μετά την συνάντηση με τον κύριο Γιούγκερ και τον κύριο Τραμπ. Είναι αυτά σύμφωνα με την τελευταία παράγραφο της μελέτης όπου κάνει το λόγο για περισσότερη διεθνή συνεργασία Ποια είναι η αξιολόγησή σας σε αυτή την μικρή συμφωνία που σύναψαν αυτοί οι μεγάλοι άνδρες. Εφτά λεπτά για να απαντήσετε στις ερωτήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε την Κίνα και το κενό εξουσίας και πώς η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να οικοδομήσει ένα βιώσιμο μέλλον ε, που να βασίζεται στην ποιοτική ανάπτυξη και όχι σε βάρος άλλων στοιχείων. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προφανώς και έχει δικό της θεματολόγιο και δικούς της στόχους βιωσιμότητας. Όμως αυτό έχει να κάνει και με τους Ευρωπαίους πολίτες. Θέλουν ε, περιβαλλοντικά κεφάλαια ε, στις ε, συμφωνίες Επομένω, δεν ε, έρχονται από το πουθενά όλα αυτά τα στοιχεία. Είδατε, υπήρχε και εκστρατεία για, το, για τη λήξη των διαπραγματεύσεων για τη συμφωνία TTIP. Πρέπει λοιπόν να γίνεται ένα screening, μια, ε, ένας έλεγχος σε ό,τι αφορά τις ε, άμεσες ξένες επενδύσεις. Εγώ δεν έχω να σας προσφέρω μεγάλες λύσεις και μεγαλόπνοα σχέδια. Έχουμε όμως μικρά λιθαράκια που μπορούμε να προσθέσουμε εδώ και βοηθούν αυτά που σας προανέφερα ε, σε ό,τι αφορά την κυβερνοασφάλεια, τις ε, κρατικές επιχορηγήσεις και το εμπορικό θεματολόγιο. Υπάρχουν λοιπόν ορισμένες χρήσιμες προτάσεις. Τώρα, κατά πόσο όλα αυτά θα συντονιστούν με το σωστό τρόπο και να παρουσιαστούν ως ένα συνεπές και συνεκτικό όραμα, αυτό είναι κάτι άλλο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι πολύμορφη, έχει ένα ευρωπαϊκό όραμα μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πρέπει να σταματήσουμε λοιπόν τις, τις διαμάχες μεταξύ κρατών μελών. Εγώ είμαι υπέρ της ε, ε ολοκλήρωσης γιατί πιστεύω ότι οδηγεί σε μεγαλύτερη επιρροή ε, και καλύτερες δυνατότητες αντιμετώπισης ε, παγκόσμιων προκλήσεων, όπως είναι η κλιματική αλλαγή. Έχουμε την ε, Συμφωνία των Περισσίνων, αλλά χωρίς τις ΗΠΑ καταραίει. Χρειαζόμαστε λοιπόν καλούς μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και στις χώρες μας. Δεύτερον, και πάλι η κοινοβουλευτική διάσκεψη κατά πόσο είναι χρήσιμος ε, μηχανισμός. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επιμένει στις ε, αρχές και αξίες της, γιατί αν αρχίσει να αλλάζει δραστικά τα πράγματα, αυτό αποσταθεροποιεί περαιτέρω την κατάσταση και δεν υπάρχει ε, μία και μόνη λύση. Όπως και στο Brexit, αυτό μάθαμε, ότι υπήρχε μόνο μία αντίδραση και ακόμα δεν έχουμε ε, καταλάβει τι ακριβώς θα γίνει. Δεν είναι ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί ε, ε, θίγει πολλούς τομείς που δεν είχαμε προβλέψει στο παρελθόν. Αν ήταν πολύ αφηρημένη η έκθεση. Εγώ είμαι δικηγόρος εμπορικού δικαίου. Με τις πρώτες με τα πρώτα προσχέδια, λοιπόν, το πρόβλημα που είχα εντοπίσει είναι ότι δεν ε, ε, ασχολούνται αρκετά με το ζήτημα του διεθνούς εμπορίου. Ξέρω λοιπόν ότι μπορεί να μην έχω καλύψει άλλα στοιχεία που έχουν να κάνουν με την Κίνα, αλλά υπάρχει ξεκάθαρη εντολή αυτή η έκθεση να αφορά και την διπλωματία και την εμπορική πολιτική. Γι' αυτό και άφησα κάποια στοιχεία εκτός. Η Ευρωπαϊκή Στρατηγική κάθε χώρα είναι πολιτικός φορέας. Ένα από τα μεγάλα ευρήματα και προβλήματα σήμερα είναι ότι η διαμόρφωση πολιτικής δεν αξιοποιεί ε, εμπεριστατωμένα επιστημονικά στοιχεία για την τεκμηρίωση των πολιτικών. Και έτσι υπάρχει ε, μία ανισομέρεια και αυτό το παρατηρούν και οι πολίτες. Καλές λοιπόν ε, οι δηλώσεις και οι μεγαλοστομίες για την διεθνική κυριαρχία και τον έλεγχο των συνόρων, αλλά στην πράξη τα πράγματα δεν έχουν πάντα την ίδια μορφή. Κάποιοι ξεχνούν επίσης ότι όταν ολοκληρώθηκε ο γύρος της Ουρουγουάης, ήταν σαφές ότι κάπου χάναμε, κάπου κερδίζαμε. Ο Τραμπ έχει ξεχάσει ότι υπήρχε μία ενιαία συλλογική προσπάθεια και αυτός τώρα προσπαθεί να την κατακαιρματίσει. Μπορεί να πάρει ένα στοιχείο και να πει «Να, ορίστε, εμείς χάνουμε εδώ». Αλλά αυτό δεν αποδίδει σωστά την ε, συνολική κατάσταση. Γιατί τελικά κάπου κέρδισε, κάπου έχασε η κάθε πλευρά και καταλήξαμε σε μία συμφωνία. Έτσι είναι οι διαπραγματεύσει, γιατί αφορούν ε, μία σειρά κλάδου και όχι μόνο έναν. 16 συν 1, Κίνα, κυβερνοασφάλεια και Βόρειος Αφρική. Εγώ ασχολούμαι με την οικοδόμηση δυναμικού ε, και στην Αφρική και αλλού και στο Αφγανιστάν. Εκεί λένε ότι δεν θέλουμε να επενδύσει η Κίνα στο Αφγανιστάν. Και στην Αφρική όμως και εκεί αλλάζει η τάση βλέπουν ότι η Κίνα έχει πολύ πιο μακροπρόθεσμο ε, πλάνο 100-150 ετών και όχι 5 και 10 πλάνο. Και η Δύση δεν σκέφτεται με αυτό το μοντέλο. Τι πρέπει να κάνουμε. Να έχουμε αυτά τα πρότυπα. Κάποιοι βέβαια Μπορούν να πούν ότι να, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλει τα ιδεολογικά της πρότυπα σε όλο τον κόσμο. Αυτά είναι τα ίδια πρότυπα που προστατεύουν χώρες από μη βιώσιμες επενδύσεις, ε, την υποβάθμιση του περιβάλλοντος ε, και της παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτά είναι τα πρώτα που χρειαζόμαστε για να λέμε να αυτό είναι που θέλουμε, αυτό είναι το επίπεδο διαβίωσης που θέλουμε και δεν πάμε παρακάτω. Και σίγουρα στην Αφρική αρχίζουν να αλλάζουν στάση ό,τι αφορά τις επενδύσεις από την Κίνα. Αν ε, είναι πια πολύ αργά, αυτό είναι κάτι άλλο. Με τον ΠΟΕ το επίτευγμα ήταν ότι βασιζόμασταν σε ένα σύνολο κανόνων υπήρχε πλέον μη, ένα διαφανές ε, σύστημα βάση κανόν και φαίνεται ότι επανερχόμαστε στο παλαιότερο μοντέλο των ε, διπλωματικών διαπραγματεύσεων με βάση την ισχύ του καθενός. Ε, και αυτό βέβαια, πιο ζημιώνεται από όλο αυτό, οι πολίτες που θέλουν να έχουν πρόσβαση στην πληροφορία και οι επιχειρήσεις που θέλουν ένα διαφανές πλαίσιο δραστηριοποίησης. Πολλά λοιπόν έχουν αλλάξει, αλλά ακόμα υπάρχει μία σειρά λόγων για τους οποίους αυτό το μοντέλο με βάση κανόνες είναι θετικό για όλους. Ε, ανεξάρτητα από πολιτικές αντιδράσεις που ακούμε σήμερα. Και σίγουρα η προσωπικότητα του Τραμπ ε, είναι αυτή που είναι πιο απρόβλεπτη σήμερα. Γιατί έχει κάποιους ευνοούμενους, κάποιους αντιπάλους, ε, κάποιοι από αυτούς αλλάζουν θέση την μέρα στην άλλη, κανείς δεν ξέρει τι θα γίνει αύριο και αυτό υποβαθμίζει ε, και υποσκάπτει ε, αυτό το σταθερό οικοδόμημα. Υπάρχουν στοιχεία που μας δείχνουν ότι αυτό δεν θα έχει θετική έκβαση στο μέλλον. Τώρα για την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα είχαμε προβλήματα στο γύρο της Δόχα αν όλοι είχαν το ίδιο θεματολόγιο. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να προβάλλει τις επιθυμίες των πολιτών της. Και αυτό μπορεί ε, να συμπεριλαμβάνει και ε, ζητήματα των ε, φίλων, των, της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ. Ανταποκρίνονται λοιπόν σε ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Και αυτό θα πρέπει να το αναγνωρίσουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι προσπαθεί να έχει τουλάχιστον ένα όραμα βιώσιμη ανάπτυξη. Δεν λέω ότι είναι τέλεια η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, για, στη χώρα μου υπήρχε πάντα ευρωσκεπτικισμός, αλλά δεν νομίζω ότι ε, λειτουργεί ισοπεδωτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπάρχει ζήτημα με τη Γεωργία παντού, αλλά και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι τα λόμπι αυτά των κρατών μελών που ασκούν πιέσει. Δεν είναι μία και μόνο Πρόκειται για μια κοινωνική αντίδραση που δηλώνει την απογοήτευσή της ε, με την παγκοσμιοποίηση. Και πρέπει να διασφαλίσουμε λοιπόν ότι δεν αυξάνονται οι ανισότητες. Και πρέπει να ακούσουμε τους πολίτες. Τι λένε λοιπόν οι πολίτες ουσιαστικά ότι πρέπει να υπάρχουν τέτοια περιβαλλοντικά ε, και εργασιακά κεφάλαια στις ε, συμφωνίες και προάσπιση των συμφερόντων τους και των δικαιωμάτων τους από τους πολιτικούς. Λοιπόν, είναι δύσκολη περίοδος, δεν υπάρχουν μεγάλες λύσεις. Από την ιστορία βλέπουμε ότι ο προστατευτισμός και οι δασμοί δεν ωφελούν μακροπρόθεσμα. Το περιβάλλον είναι σημαντικό καθώς και η μετανάστευση παγκοσμίω και ε, η συγκέντρωση κυριαρχίας ενισχύει τις θέσεις εμμονωμένων κρατών μελών. Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστώ όλους όσοι συμμετείχατε σε αυτή, στην εκπόνηση αυτής της ε, μελέτης. Ο Bob έλεγε «Times are changing», αλλάζουν ε, οι καιροί. Ωραία, φτάνουμε στο τέλος. Καλό βράδυ.